πλέον. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε παρατηρήσεις ε, επ' αυτών. Όχι από ό,τι βλέπω. Άρα εγκρίνουν τα πρακτικά και περνάμε στην ψηφοφορία. Και ξεκινάμε με, τις, ε, με κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκασπάρη, διαδικαστικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε κύριε Βίλαντ, αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση το άρθρο 22.4 του κανονισμού μας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο προς τα έξω. Οι θέσεις του Κοινοβουλίου καθορίζονται ε, από κοινού σε ψηφοφορίες, άλλες από αυτές κερδίζουμε, σε άλλες χάνουμε, αλλά ως δημοκράτες δεχόμαστε πάντα ε, τα αποτελέσματα. Εχθές ο κύριος Σούλτς εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο, στη συνάντηση κορυφής και για άλλη μια φορά εξέφρασε τις προσωπικές του απόψεις και όχι τις δικές μας. Παράδειγμα, το Κοινοβουλίο τοποθετήθηκε στο θέμα της προστασίας των επενδύσεων ε, στην έκθεση Γκαντία Ρίφ ε, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία και επίσης ε, και το ψήφισμα Μορέρα και αυτό στηρίχθηκε. Το να μην λαμβάνει υπόψη το ίδιο ο πρόεδρός μας τα ψηφίσματά μας, τότε δεν χρειάζεται να εκπλήσουμε το ότι δεν μα λαμβάνει υπόψη σοβαρά ούτε και άλλοι όπω το Συμβούλιο Υπουργών. Επειδή έχει συμβεί αυτό επανειλημμένα, παρακαλούμε όλοι ο πρόεδρος και οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου να διασφαλίζουν σε επίσημες εκδηλώσεις να εκφράζεται και η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κασπάρη. Θα το λάβουμε υπόψη. Καταγράφεται ο κύριο Μπιούτικοφερ, χωρί μικρόφωνο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο να συσταθεί η Επιτροπή για την εξέταση της ορθής εκπροσώπησης των αποφάσεων του Κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο. 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες 24 ώρο, πρέπει μια Επιτροπή να παρακολουθεί τι πράττει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Βιουτικόφερ, Ψηφοφορίες. Κοινό ψήφισμα. Έξι ομάδων για το Σουδάν. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος για την Αίγυπτο. Έξι ομάδων. Η έκτη παράγραφος σε δύο Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τιολογική σκέψη 1 αρχικό τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Q σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Προχωρώ στην ψηφοφορία του ψηφίσματος του σχετικού με την Ιγυρία που έχουν καταθέσει έξι ομάδες και πάλι και έχουμε μία πρόταση μια τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Όπω τροποποιήθηκε το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά υπέρ. ε, ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται επίση. Κυρίε και κύριοι, έχω μια ανακοίνωση για τις προτάσεις των διασκέψεων των Προέδρων για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, άρα τα μέλη εκλέγονται όπως ε, έχουν προταθεί από τη διασκέψη των Προέδρων και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία, ένα κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων και των συναδέλφων Ματσερόνη και Γκρικούλε. Τροπολογία υπαριθμών 6 καταρχάς υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 με μια προφορική τροπολογία από τον συνάδελφο Σάριους Βόλσκι. Έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Θα θέλαμε να προσθέσουμε την εξής φράση, κύριε Πρόεδρε. Καλοί αντάρτες και μισθοφόρους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και να μην χρησιμοποιούν τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, άρα ψηφίστε με αυτή την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 χωριστά σε τρία τμήματα. Ονομαστικά κάθε φορά. Πρώτο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. εγκρίθηκε τρίτο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται τροπολογία νέα ονομαστικά άρχεται ψήφισαν όλοι πέρας Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Αρχικό κείμενο καλύπτεται ως εκ τούτου από την τροπολογία. Παράγραφος 12 με τον κύριο Σάρους Βόλ προφορική τροπολογία. Στο τέλος του κειμένου να βάλουμε τις εξής λέξεις. Καλή κάθε πλευρά να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσοδέψει τους αμάχους και να εξασφαλίσει την ε, ε, διαβίβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. Κύριε Σάρος η τροπολογία 9 έχει εγκριθεί και ως εκ τούτου έχει καταπέσει το άρθρο της παραγράφου 8. Εσείς κάνετε αναφορά σε τροπολογία προφορική για την παράγραφο υπαριθμών 8, η οποία όμω πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και τώρα έχουμε περάσει στην παράγραφο 12. προφορική τροπολογία για την παραγράφο 12 ζήτησα να μου εκθέσετε, όχι για την 8. Paragraph 8 was Έχει καταπέσει η παράγραφος 8. Η 8 έχει καταπέσει. Θέλετε να καταθέσετε προφορική τροπολογία για την 12 νέου. Ου. Καλώς. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την παράγραφο 12. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 2 επί της παραγράφου 12, ονομαστικά αρχίζει. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. Απερίφθη. Τροπολογία 10 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 11 ονομαστικά. Αλλά με προφορική τροπολογία του κυρίου Σάιρους Βόλσκι. Στο τέλος και μετά τη λέξη ρητορική να βάλουμε και τις λέξεις περιλαμβανομένες της ουσίας και μετά να συνεχίσουμε μπορεί να επιδεινώσει της ε, ε, τη σύγκρουση. Υπάρχουν αντιρρήσει προ την κατάθεση προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν ονομαστικά την τροπολογία 11 με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. τρία τμήματα. Πρώτο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Λέει ο πρόεδρος. Το υπαριθμόν 2 επαληθεύεται παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι παντές. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πάλι με προφορική τροπολογία του κ. Σάριου Βόλσκη. Είναι μια προφορική τροπολογία στην προφορική τροπολογία των Πρασίνων. Ο κ. Σαρσβόλ και προτείνω σε αυτή την τροπολογία να απαλείψουμε στον τρίτο στίχο τη λέξη και με την κυβέρνηση τη Ουγγαρική κυβέρνηση να υπογράψει με τη Ρωσία αυτή την συμφωνία για την υπηρετική ενέργεια. Οπότε να απαλληφθεί αυτό και να γίνει απάλληψη στου στίχου 3 και 4 και να υπογράψει η Ουγγρική κυβέρνηση αυτή την... Αυτό, να απαλληφθεί αυτό που αναφέρει η Ουγγρική κυβέρνηση και την τη συμφωνία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Τουλάχιστον 40 συνάδελφοι, ως εκ τούτου ψηφίζουμε μόνο την αρχική μορφή της τροπολογίας. Αρχής ψηφοφορία για την 5. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. Απερίφθη 7 κατά άποχες εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ αρχίζει. Ψήφισετε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ε, στα ψηφίσματα ε, θέσεις απασχόληση για τους νέους έχουμε πρώτες ψηφίσματος από τέσσερις πολιτικές ομάδες ή εννέα. Σε ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές γκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Τροπολογία 4 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ε, τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 11 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 16, αρχικό ε, κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται λάθος ο πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα πρωτοτμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μισό λεπτό. Ε, παληθεύουμε. Ψηφίζουμε. Ε, ψηφίσατε όλοι έκλειση ψηφοφορία. Κοιτάξτε, παρότι πολλές αποχές εγκρίνεται οριακά, λέει ο πρόεδρος. Η τροπολογία 7, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 42 αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα, όλα μονομαστική ψηφορία, πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 43 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 44 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 8, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 45. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Διαδικαστικό παρακαλώ θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια προφορική επεξίσχερη με αυτό η οποία έγινε αποδεκτή προηγουμένως για το 45 όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης δικής των εργαζομένων εκεί που λέμε κατηρτισμένοι με δεξιότητες πρόεδρος συγγνώμη επεξήγηση ή προφορική τροπολογία προφορική δήλωση για την ψηφορία επεξήγηση που είναι μετά τι ψηφορίε. ευχαριστώ Πάμε στην 44. Ε, ε, Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Μισό λεπτό ξανά. Υπέρ. Εντάξει, εγκρίθηκε. Παρακαλώ, συνάδελφε, μου επιτρέπετε να κάνω μία πρόταση. Ξέρετε, εγώ νέο είμαι εδώ, παρόλα αυτά όμω έχω κοινοβουλευτική εμπειρία. Μην μου θυμώνετε, αλλά θα ήταν καλό να έχουμε τουλάχιστον το χρόνο ανάμεσα στο υπέρ, κατά και εγκρίνεται να σηκώνουμε το χέρι μα. λέτε τόσο γρήγορα ούτε χέρι δεν προλαβαίνουμε να σηκώσουμε. Λυπάμαι, αλλά πάτε πολύ γρήγορα, πρόεδρε. Πρόεδρος, συνάδελφε, Ευχαριστώ ε, να κάνω πιο αργά, αλλά θα δείτε ότι μερικοί συνάδελφοι, αν ε, πάμε αργά, θα αρχίσουν να φεύγουν. Όλοι περιμένουν να φύγουν, τους περιμένουν τα αεροπλάνα και κάνουμε το ρυθμό που είχε καθιερωθεί στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και Γι' αυτό το λόγο έχετε και τους καταλόγους μπροστά σας. Οι συνεργάτες σας σας έχουν προετοιμάσει τους καταλόγους ψηφοφορίας. Γι' αυτό το λόγο. Μισό λεπτό. Μετά το 14 έρχεται η τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μετά το ε, ΚΑ, ε, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ, το εκτιμώντας ΚΑ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος, ε, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για την κατάσταση στο ΙΚΡΑΚ. Έχουμε κοινό ψηφίσμα από πέντε πολιτικές ομάδες. Καταρχήν η τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του έχω και μία ε, προφορική τροπολογία της συναντέλφου κυρίας Γκόμες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα εδώ, γιατί μιλάμε για τις 15 Ιουλίου, όχι 14. Στο, στην έκτη παράγραφο. Τεχνική διόρθωση. Καλώς ορίζει την εκλογή του νέου Προέδρου του Ιρακίνου ε, Κοινοβουλίου στις 14 Ιουλίου γράφει. Στο κείμενο πρέπει να είναι 15. Μια τεχνική προσαρμογή ζητάω. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Θα το ελέγξουμε και αναλόγως θα το διορθώσουμε. Τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα πρόταση ψηφίσματος για την κλιμάκωση βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, κοινό ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων, ε, τροπολογία 6 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, η 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, η 2 ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 1 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τρία ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μετά το εκτιμώντας G, ε, το 5, ψηφίζουμε παρακαλώ για το 5. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα ε, το ψήφισμα στο σύνολό του. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Και τώρα περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος ε, με θέμα έγκλημα της επίθεσης. Ε, έχουμε ε, μία πρόταση από μία πολιτική ομάδα, του συντηρητικού κυβερνητές, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στο κοινό, κοινή πρόταση ψηφίσματο πέντε πολιτικών ομάδων και έχουμε μόνο μία ψηφοφορία σχετικά με το εκτιμώντα F αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την ψηφοφορία για το ψήφισμα ως δεν έχει τροποποιηθεί υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και έχω και μία ανακοίνωση να σας κάνω. Ο κύριος Κάλλος Χιμένες Φιλαρέχο μου ανακοίνωσε την ε, παρέτησή του ε, από την 1η Αυγούστου του 2014. Και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο ανακοινώνει ότι όσον αφορά την ε, θέση αυτή του κυρίου Κάλλος Χιμένης Μιναρέχο η θέση αυτή χειρεύει και θα ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλλον. Και όσοι ταξιδεύετε σας εύχομαι